Thank you, colleagues. Um, Ευχαριστώ συνάδελφοι και όπως ε, ξέρετε είναι στενά τα χρονικά περιθώρια σήμερα γιατί έχουμε και την επόμενη ακρόαση. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα το δούμε τώρα. Έχουμε καθυστερήσει κιόλας λίγο να προχωρήσω γιατί είναι εδώ και ο εισηγητής ε, στο σημείο 4 λοιπόν έχουμε τον ε, κύριο Νάντζη για τα ελάχιστα πρότυπα για τις ε, μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νάντζη και συνάδελφοι. Αν θέλετε να φύγετε από την αίθουσα, παρακαλώ τουλάχιστον να κάνετε ησυχία. Παρακαλώ κύριε Νάντζη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Colleagues, uh, please leave as quietly Συνάδελφοι, παρακαλώ, αν μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα ήσυχα. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε Νάτζη, δεν μπορείτε να περιμένετε άλλο, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να σας παρουσιάσω το σχέδιο της έκθεσης της πρωτοβουλίας για τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους κοιόντες για την βοήθειά τους, ε, τα μέλη της ομάδος για τα δικαιώματα για τις μειονότητες, την τεράστια υποστήριξη από πλευράς του Πρόεδρου. Σας ευχαριστώ. Το Γραφείο για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα στην Βιέννη, το ECMI, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα θέματα των μειονοτήτων και πολλές μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, όλους τους εμπειρογνώμονες και το Η προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητων αποτελεί μια προστασία όλης της κοινωνίας. Ε, αποτρέπει λοιπόν συγκρούσεις που οδηγούν σε τριβές και συγκρούσεις. Γι' αυτό λοιπόν είμαι περήφανος που εκπρόσωπο την ομάδα μας για να καταδείξουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον με την προστασία των μειονοτήτων όλων των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο λοιπόν της έκθεσης βασίζεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής, ε, του χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα καρτία της Κοπενχάγης και τα έγγραφα του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες στον Ευρωπαϊκό Χάρτη, για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες που έχουν προσυπογράψει σε πολλά κράτη-μέλη. Το κείμενο λοιπόν ασχολείται με τρεις πυλώνες των εθνικών ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων κατάρτιση, πολιτισμός και δικαιώματα σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, βάσει και της αναλογικότητας και της επικουρικότητας εξαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα και τα θέματα αυτοδιάθεση και αυτοδιακυβέρνησης, τοπική αυτοδιοίκησης. Ε, αυτό επαφείται στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη το καθορίζουν. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για την πολιτική συμφωνία για το θέμα αυτό. Το ψήφισμα για την προστασία των μηνοτήτων, λοιπόν, και οι πολιτικές κατά των διακρίσεων παρουσιάστηκαν από τον ε, πρόεδρο, τον κύριο Κλοντ Μωράης. Από τα κριτήρια της Κοπεχάγης έχει υπάρξει μια συνθήκη, αλλά δεν υπάρχει δέσμευση ότι φατηρούνται τα κριτήρια της Κοπεχάγης μετά την ε, προσχώρηση στην Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να πάμε και παραπέρα. Να υπάρξει οδηγία για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειονοτήτε λοιπόν αυτέ. Ε, θα πρέπει να γνωρίζονται ότι και αυτό να αποτελέσει όρο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα υπενθυμίσω ότι στο πακέτο πρωτοβουλίας ε, για τα δικαιώματα των τον φέτο. Συλλέχτηκαν 1,3 εκατομμύρια υπογραφέ για την προστασία των ατόμων που εντάσσονται σε πολιτισμικέ και γλωσσικέ μειονότητε, προκειμένου να ενισχυθεί και η πολιτισμική ποικιλία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι πρόκειτο για τι ίδιε δραστηριότητε όπω η έκθεση αυτή ξεχωριστή πρωτοβουλία. Το 2013 ξεκίνησε και στην τελική ανάλυση το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέρσι το 2017 αποφάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να λάβει υπόψη την πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τις αστυνικές και γλωσσικές ε, πρωτοβουλίε. Πρωτοβουλία των πολιτών περιλαμβάνει 1,3 εκατομμύρια υπογραφέ. Αλλά ξέρουμε ότι οι εθνικέ μειονότητε ε, και οι γενικότερε μειονότητε αφορούν 14 εκατομμύρια ανθρώπου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το FRA συμπεραίνει ότι όταν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνολική δικαιοδοσία για την νομοθεσία, μπορεί να αποφασίσει για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τα άτομα που εντάσσονται σε μια ομάδα μειονότητα. Έχουμε και πολύ συγκεκριμένα έγγραφα από το Σύμβολο τη Ευρώπη. Ψήφισμα 1985 του 2014, το οποίο απαριθμεί τι λεπτομερεί ανάγκε των αστυνοτικών μειονοτήτων και επίση τονίζει ότι υπάρχουν πολλέ καλέ πρακτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, Χολστάιν, Φιλανδία. Αυστρία, στην Ιταλία, στο Τυρόλο. Αυτέ οι βέλτιστες πρακτικές λοιπόν θα πρέπει να διανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών. Επίση, αναφέρονται ειδικές ανάγκε των μειονοτήτων, για παράδειγμα, δυνατότητε εκπαίδευση σε, σε μειονοτικές γλώσσες και στην Ήπεθρο και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στην ε, γλώσσα μειονότητας δεν θα πρέπει να τύχει το θέμα των χρημάτων για τη διαχείριση μικρών σχολείων. Το θέμα είναι το δικαίωμα να έχει κανείς εκπαίδευση στην μητρική του γλώσσα και ως λύση για αυτές τις ειδικέ ανάγκες η έκθεση αυτή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει να προβεί σε νομοθετική πρόταση για ελάχιστα πρότυπα για τις μηνότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή για τις τροπολογίες, αν θέλετε να καταθέσετε προθεσμία μέχρι 21 Ιουνίου. 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Νάγκη. Είπα στους συναδελφούς ότι το προγραμματίσαμε αυτό μαζί ε, τώρα και πιεζόμαστε. Το κάναμε σαν μεταξύ των δύο ακροάσεων. Μετά έχουμε για το Facebook την Oxford Analytica την ακροστρό. Ε, έχουμε τους σχεδόν ηγητές. Κυρία Σπινέλη, κυρία Γιούροβα, Γιουρόκα τέλο πάντων. Πάρκο να είστε σύντομοι γιατί δεν γίνεται αλλιώς Ρίξτε μια ματιά στο, στο πρόγραμμά μας. Πιο σφιχτό δεν γίνεται. Τρία λεπτά. Εντάξει. Μα θα το ξανασυζητήσουμε. Με πιο καλές συνθήκες. Σόραγε. Εσείς η σκιώδης για τους σοσιαλδημοκράτες. Έγινε η πρώτη των σκιωδών περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ήρθαν οι διάφορες σκιώδης ηγητές, ήρθε ο κύριος ε, ε, Νάγκη, ήταν πολύ αξιόλογη αυτή η συνάντηση και Καταλαβαίνω γιατί στείλει την προσοχή του στους τρεις πυλώνες. Όμως είναι σημαντικό να καλύψουμε και άλλα θέματα που αφορούν τις εθνοτικές μειονότητες. Ε, τα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά τους. Οπότε πρέπει να προσθέσουμε και ε, άλλα κεφάλαια. Να σας διαβάσω απλώς, απλώς τους ε, τίτλους και όχι το περιεχόμενο σεβασμός και προστασία ταυτότητας. Ε, δικαιώματα των πολιτών, πολιτικά δικαιώματα, καταπολέμηση ευρωτικών μορφών, δυσμενούς ε, διάκρισης και περιθυροποίησης. Αυτό περιέχεται και σε ψήφινα του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίσης ε, ενεργή, ουσιώδης συμμετοχή. Επίσης κάποιες σκέψεις για τα ήδη παρόντα στο κείμενο. Δηλαδή, είναι σημαντικό η ιστορία της μειονότητας να είναι ύλη του σχολείου, να διδάσκεται για τους τσιγκάνους, για την Ισλαμοφοβία και λοιπά. Επίσης ε, κάποιες επέτειοι, γιορτές τους να τιμούνται από το κράτος. Επίσης νομοθετική κατοχήρωση κάποιων πολιτιστικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και είμαι βέβαιο ότι συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά κυρία Σπινέλη πριν την κυρία Γιούροκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Μαρίνα Αλμπιόλ ζητεί να την συμπαθούμε που δεν μπόρεσε να παραστεί να σας τα πω εκ μέρους της. Πρώτα πρώτα ευχαριστεί τον εισηγητή, θεωρεί ότι είναι καλή αφετηρία το κείμενό του. Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων θα πρέπει να γίνει με τρόπο δυναμικό, θετικό, να σεβαστούμε τη διαίρεση των εξουσιών ή μάλλον την κατονομία αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και ένωσης υπάρχει σφαιρική προσέγγιση από το κοινωτικό δίκαιο όταν έχουμε κάποιες θεσμικές εκφράσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και δυσμενούς διάκριση. Η κυρία Αλμπιόν θέλει επομένως να δούμε τα διαρθρωτικά, τα συστημικά θέματα αυτών των δυσμενών φαινομένων που θίγουν τις μειονότητες. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε επίπεδο τα όργανα ε, να ενεργούν ε, δραστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων μειονοτήτων και να τονίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει ορισμός της μειονότητας. Αυτό όμως να μην είναι φραγμός στην ανάληψη δράσης όπου θεωρούμε ότι συντρέχει περίπτωση δυσμενών διακρίσεων. Και η αποφυγή των διακρίσεων είναι η βασική προσέγγιση για την προστασία αυτών των ανθρώπων το να υλοποιηθεί είναι βασικό, λέει η κυρία Αλμπιόλ. Οπότε τα εγκλήματα μίσους, ε, ο λόγος μίσους θα πρέπει να καταπολεμηθεί και με πολιτικές να φαραγγίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τώρα όσον αφορά τα γλωσσικά, όσον αφορά την προσβασιμότητα στις κρατικές υπηρεσίες σε όλες τις γλώσσες, αυτό να είναι εγγυημένο να μην είναι η γλώσσα των διοικητικών διαδικασιών λόγος περιθωριοποίησης. Ε, έχουμε τώρα το ψήφισμα τη 25η Δεκάτου του 2017 για κάποια βασικά ζητήματα όσον αφορά την γενική ένταξη των Ρωμά στην Ένωση. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η τσιγκανοφοβία. κύριε Αλμπιόλ θεωρεί ότι αυτά όλα που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι κάτι που αξίζει να λάβουμε υπόψη για την έκθεση. Κυρία Γιώργα, έχει το λόγο, αλλά κάνουμε και ένα διάλειμμα πριν την ε, ακρόαση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον εισηγητή, να πάει το έγγραφο αυτό με όσο το δυνατόν πιο καλά αποτελέσματα για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και για την ε, προσήλωση και στράτευση και πλευρά των σοσιαλιστών για τις ε, διακρίσεις και την ομοθεσία. Όταν έχουμε νομική βάση για το έγγραφο, με σαφή και δυνατότητα να παρακολουθούμε τα επιτεύγματα και την πρόοδο, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να χάσουμε χρόνο σε κενές υποσχέσεις από πλευρά της Επιτροπής. Θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ας μιλήσουμε λοιπόν κατευθείαν για κυρώσεις. Το έγγραφό σας βέβαια είναι σαφώς ξεκάθαρο ενισχύει την κοινωνία των πολιτών Επιτρέπει δηλαδή στον πολίτη, στον να υψώσει τη φωνή του, δεν θα τον φημώνει κανείς, δεν θα εκφράζει κανείς τον πολίτη στη θέση του. Γιατί πρέπει πράγματι όποιος είναι επί τόπου καταλαβαίνει την κατάσταση, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς άλλος για λογαριασμό τους. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμά σας. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με, όλες τις, με όλα τα θέματα. Οι μειονότητες όντως είναι φτωχές. Ας μην μιλούμε λοιπόν μόνο για δικαιώματα, Α μην εξαντλούμε τη συζήτηση στα δικαιώματα, αλλά α κάνουμε πράγματα και για την οικονομική ενσωμάτωση, γιατί μιλούμε για διπλή και τριπλή πολλέ φορέ. Ε, ε, διπλό και τριπλό αποκλεισμό από την κοινωνία των ανθρώπων αυτών. Παρακαλώ, κύριος Νάγκη. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Οπωσδήποτε Θα αναφερθούμε και στις ε, μειονότητες. Θα έχουμε μια καλή, πιστεύω, και ομαλή συνεργασία με την υποστήριξη και των συναδελφών από τις ε, άλλες ομάδες. Ευχαριστώ κύριε Νάγκη. «21 Ιουνίου προθεσμία και τώρα 10 λεπτά διακοπή πριν από την ακρόαση για το Facebook που θα ξεκινήσει ακριβώς στις 17.30. Δεν ξέρω αν έχετε και σαν και για μια μικρή διακοπή όπως εγώ. Περνάμε λοιπόν ακριβώς 17.30 στην ακρόαση για την Cambridge Analytica και το Facebook.